κατάλαβα νομίζω και αιτιολόγησε με βάση το άρθρο 138 απλοποιημένη διαδικασία για τέσσερις εκθέσεις. Πρώτα η έκθεση του κυρίου Νίκου Λέσχου προφορική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Να περάσουμε στην έκθεση τάιν για το δίκαιο που πρέπει ε, να ε, ισχύει για τις καταχωρημένες ε, συμβιώσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Επίσης, έκθεση Time, η επόμενη έκθεση. Για, τις, για το εφαρμοστέο δίκαιο, για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το γαμικό δίκαιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος, έκθεση Κρέμα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών και για την μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης και κινητικότητα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κύριε Λίζε, είστε πολύ αθλητικός. Ψηφίσατε. Ωραία, πέρασε. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα στην έκθεση της κυρίας Αντωνέσκου. Α, ήρθε ο συγητής. Καλώς ήρθατε. Κύριε Κράμερ, εγκρίθηκε το μεταξύ έκθεσή σας. Υποθέτω ότι κολλήσατε στο ασανσέρ. Βεβαίως. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση Αντωνέσκου για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο κατά ποινικέ διαδικασίες και δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την ε, ούτως τροποποιημένη πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία η οποία και άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται συγχαίρω την κυρία Αντωνέσκου Τώρα περνάμε στην έκθεση του συνάδελφου Σάντσεθ Πρεσέδο για συμβάσεις πίστοσης για ακίνητα κατοικίες. Ε, ψηφίζουμε στο μπλοκ 1 τροπολογία 117. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο μπλοκ 1 οι 1 62 καταπίπτουν. Ε, τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Κύριε Σάντσεφ Εθπρεσέδο, ζητήσατε το λόγο πριν την ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Παρακαλώ. Μετά του τριμερείς διαλόγους, το μόνο εκρεμές ε, θέμα είναι ένα τεχνικό που αφορά τη διαδικασία μετάθεσης στην εσωτερική νομοθεσία. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποσαφινιστεί και την εκφράσαμε με σαφήνεια. Ε, και μετά από συνεννόηση με τους ε, εισηγητές και με βάση του, τους, τη σύσταση των συντονιστών, προτείνω με βάση το 52 2 του κανονισμού να αναβληθεί η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η ε, εκκρεμούσα διαπραγμάτευση. Ωραία, ο εισηγητή θέλει ε, αναβολή με βάση το 57.2 του κανονισμού από ό,τι κατάλαβα. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Οπότε αναβάλλεται η τελική ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην έκθεση της συναδέλφου Μακάθη. Επιστευτικές προφορίες και πράξη χειραγώγησης αγοράς. Ε, να περάσουμε στην τροπολογία 2. Κατά τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά άποχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε το μπλοκ 2 και η τροπολογία 1 καταφύπτουν. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαίρω την κυρία Μακάρθη. Τώρα έκθεση Γκρομπάρτσικ. Τροποποίηση του κανονισμού 287-2005 του Συμβουλίου. Τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων στην Βαλτική, στο Μπέλτ και στο Σάουντ. Τροπολογίες 1 έως 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος η οποία και άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαίρω τον κύριο Γκρομπάρτσικ. Και τώρα στην έκθεση του πρώην Προέδρου συναδέλφου Μπούζεκ για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ψηφίζουμε το άρθρο 3 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Λοιπόν, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται το 3. Άρθρο 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 40, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 44 του αρχικού κειμένου, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες ε, θεωρώ ότι απορρίπτεται εντάξει καλά ας ελέγξουμε άρχεται δεύτερο τμήμα του 59 της παραγράφου 59 πέρας ναι έχει απορριφθεί Παράγραφος 65. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα συνολικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγχαίρω τον συνάδελφο Μπούζεκ τώρα έκθεση της συναδέλφου Κλέβα Κέκους για την εφαρμογή και αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στα πλαίσια της πολιτικής για τη συνοχή το 9 παράγραφος 9 Πρώτο τμήμα. Σε τρία τμήματα την ψηφίσουμε. Υπέρ του πρώτου, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 55 όχι, όχι, ήταν σαφέ, ήταν σαφέ. Παρακαλώ, 55 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 57, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, το ψήφισμα ε, ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Κλέβα. Τώρα, έκθεση του συναδέλφου Μιλάνα, ε, ο οποίος θέλει το λόγο πριν από την ψηφοφορία, ως εισηγητής. Πού είστε, συνάδελφε Μιλάνα, παρακαλώ. μία μικρή τεχνική διόρθωση. Η έκθεση συνετάχθη πριν από την 1η Ιουλίου και η Κροατία αναφέρεται ότι βρίσκεται στην πορεία της ένταξης ενώ θα πρέπει να διορθωθεί βέβαια διότι είναι πληρέστατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Οι υπηρεσίες ah, μου είπαν κύριε Μιλάνα ότι ε, θα διορθωθεί σε όλες τι ε, μεταφράσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παράγραφος 4. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε. Ε, καλά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά. Παράγραφος 23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συγχαίρω τον κύριο Μιλάνο. Τώρα περνάμε στην έκθεση τη συναδέλφου Ντελάνγκε για περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ καλά. Υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση. Απόπειρα είπε γερμανικά ο πρόεδρο πριν διορθώσει πρόταση. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι. Ε, συγγνώμη, μία απόπειρα, όχι, μία εναλλακτική ε, από τη σοσιαλιστική ομάδα. Λοιπόν, για αυτήν θα ψηφίσουμε ονομαστικό Άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. Α, η απόπειρα επετεύχθη. Οπότε το κείμενο της Επιτροπής καταπίπτει, διότι ε, ε, πέρασε το ψήφισμα των σοσιαλιστών. Οπότε, και τώρα περνάμε στην καλύτερη έκθεση της ημέρας. Συνάδελφος Φόξ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Επιγραμμικός. Μου είπε ότι έχει ήδη στοιχηματίσει για το πώς θα ε, πάει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα την παράγραφο 2 του αρχικού κειμένου. Δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στο αρχικό κείμενο. Παράγραφος 5 πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Α, καλά. Μα ήταν σαφές. Σας παρακαλώ. Καλά, καλά. Ωραία. Α, καλά, ωραία, εγκρίθηκε, ωραία. Λοιπόν, παράγραφος 19, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Καλά, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Δεύτερο τμήμα, 19, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Ε, εγκρίθηκε, ε. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα κάτι τη γνώμη μου θα είναι ίδιος ο σχετισμός. Παρ' όλα αυτά θέλετε να ελέγξουμε. Καλά, το τρίτο τμήμα. Ωραία, ωραία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 28. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Έγκρινεται. 702. Ονομαστική για την παράγραφο 29 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται επίσης. Τώρα, παράγραφος 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εδώ η αριστερά φαίνεται ότι έχει κουραστεί και δεν μπορεί να σηκώνει το χέρι της. Όχι, όχι όπως πάντα. Σήμερα μόνο το παρατηρώ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 64 ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Ονομαστική για το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Φόξ. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε έναν διορισμό σύμφωνη, σύντομη πληροφόρηση, διορισμός του Λίτζι Μπερλιγκουέρ ως μέλους του άρθρου 255 της Συνθήκης για την Εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Επιτροπή που συνίσταται με βάση αυτό το άρθρο. Λοιπόν, έχει ανάψει ο, ο μπλε φωτισμός, μπορείτε να ψηφίσετε ναι, όχι, αποχή, αλλά δεν θα φανεί πώς ψηφίζετε. Είναι μυστική ψηφοφορία. Διορισμός του κυρίου Μπερλιγκουέν με βάση το άρθρο 2, 69 ε, του κανονισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ο κύριος Μπερλιγκουέρ εκλέγεται και τον συγχαίρω. Και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου όπου θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Μπλάζα.